Δεν ζήτησα τώρα να μιλήσω. Ίσως ε, υπάρχει κάποιο λάθος, κάποια σύγχυση. Δεν ήθελα εγώ, δεν ζήτησα το λόγο. Καλώς. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να τελειώσουμε τις παρεμβάσεις ε, ενός λεπτού και το επόμενο θέμα μας ε, είναι η έκθεση του κυρίου Σβένσον η προώθηση της ανάπτυξης μέσω εμπορικών συναλλαγών. Ο κύριος Σβένσον είναι ο πρώτος ομιλητής. Το διεθνέ εμπόριο παίζει ένα σημαντικό ρόλο για τις αναπτυσσόμενε χώρε. Νομίζω ότι αυτό είναι προφανές και συμφωνούμε όλοι γι' αυτό. Και γνωρίζουμε ότι τα πλανητήματα της παγκοσμιοποίηση μπορούν να ωφελήσουν τις αναπτυσσόμενε χώρε και τι έχουν ωφελήσει πράγματι. Και αυτή είναι η αποστολή μα, αλλά και η ευθύνη μα. να φροντίσουμε τους ώστε να συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά βεβαίω υπάρχουν και κίνδυνοι από την άλλη και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει πιο ολοκληρωμένο διεθνές εμπόριο ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν αυτοί οι κίνδυνοι. Εάν υπάρχει ελεύθερο εμπόριο, ο βασικός στόχος θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών. Καμιά φορά το εμπόριο και η βοήθεια για το εμπόριο είναι, εμφανίζονται ως αντιφατικές θα πρέπει το εμβόλιο να μπορεί να βοηθήσει τις χώρες αυτές για την ανάπτυξη και θα πρέπει αυτά τα δύο να συμπορεύονται. Άρα λοιπόν οι δύο αυτές προοπτικές θα πρέπει να συμβαδίζουν και να βελτιωθεί η εμπορική δυνατότητα των φτωχών χωρών, ε, θεωρώντας ότι η ανάπτυξή τους είναι απολύτως ε, αναγκαία. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι όλα αυτά σχετίζονται με την εξασφάλιση ενός ειρηνικού μέλλοντος. Και θα πρέπει να δούμε ότι οι εμπορικές σχέσεις με τις αναπτυσσόμενες χώρες τελικά προϋποθέτουν μια διαφορετική στάση από τη δική μας πλευρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ότι όταν υπάρχουν ισότιμοι εταίροι. Θα πρέπει να δούμε ότι αυτές οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν θα πρέπει να παραμείνουν εξαρτημένες από τις πρώτες ύλε και τους φυσικούς πόρους. Θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι θα πρέπει να γίνουν ανταγωνιστικές σε μια ισότιμη βάση ανταγωνιστικές σε σχέση με την Ευρώπη. Γι' αυτό συχνά το παραγνωρίζουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί βεβαίως θέλουμε να προστατεύσουμε τα συμφέροντα της δικής μας ε, βιομηχανίας. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να τονίσω το πόσο σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να υπερασπίσουμε, να επιδείξουμε ελεγγύη σε μια ε, πρακτική μορφή, για παράδειγμα τις εμπορικές σχέσεις και επίσης θα πρέπει να υπεραπιστούμε και τα ανθρώπινα δικαιώματα, να εξαλειφθεί η παιδική εργασία σε όλα τα μέρη του πλανήτη. Και επίσης θα πρέπει το εμπόριο να αποβεί γεργετικό για το σύνολο του πληθυσμού στο μέτρο του δυνατού δεν θα πρέπει να είναι μόνο εις όφελος των ανθρώπων στις αστικές ε, περιοχές, αλλά θα πρέπει να ωφελεί και τους κατοίκους της υπαίθρου, τις γυναίκες και τα παιδιά για παράδειγμα, που πολλές φορές χάσουν ειδικέ μορφές βοήθειας και μια ειδικότερη υποστήριξη, ιδιαίτερα όσον αφορά την πολιτική του εμπορίου. Θα ήθελα να αναφέρω μια, την ανάγκη μιας πολιτικής για την ανάπτυξη για να καταλήξω. Εμείς οι ίδιοι έχουμε δεσμευθεί όλες οι πολιτικές, η Αλία, η Γεωργία κλπ. θα πρέπει να συμβάλλει σε μια πραγματική ανάπτυξη σε ολόκληρο τον κόσμο. Και παρακαλώ να μην το παραμελούμε στην ε, πρακτική μας, καθημερινή μας ε, εργασία. Και απλώς να το αναφέρομαι μόνο όταν ε, υποβάλλεται κάποια έκθεση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ερχόμαστε στη διαδικασία Catch the Eye. Η πρώτη ομιλήτρια είναι η κυρία Μπασέσκο. Η κοινή εμπορική πολιτική είναι ένα μέσο το οποίο είναι, πλέον, είναι ωφέλιμο τόσο για τα κρατημέλη όσο και για τους εταίρους της Ένωσης. Εμπορικέ συναλλαγές με λιγότερο αναπτυγμένες χώρες ενθαρρύνουν την διαφοροποίηση των οικονομιών αυτών των χωρών και την ένταξή τους στην παγκόσμια αγορά. Γι' αυτό θα πρέπει να αποφεύγουμε τους περιορισμούς που στρεβλώνουν το εμπόριο, ώστε να επιτρέψουμε στις στοχότερες χώρες να χρησιμοποιήσουν το ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα. Η βοήθεια για το εμπόριο θα πρέπει να βοηθήσει τις ευνοψόμενες χώρες και τις προσπάθειές τους να προωθήσουν το τοπικό εμπόριο. Ταυτόχρονα πιστεύω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να βοηθηθούν οι ξένες άμεσες επενδύσεις γιατί είναι ένα σημαντικός παράγοντας για βιώσιμο πλούτο, αναπτύσσουν το επιχειρηματικό πνεύμα, τη τεχνολογία και δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Γι' αυτό είναι ουσιώδης για την ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Νικολέσκου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για την εργασία του η έκθεση όμως νομίζω ότι είναι υπερβολική σε κάποια θέματα, τα οποία ελπίζω να τα αντιμετωπίσουμε αύριο. Συζητεί για την ε, αρνητική επίδραση της Γεωργίας στην ανάπτυξη. Η Γεωργία ήδη έχει περικοπεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και χρειάζεται μεγαλύτερη σύνεση όταν μιλάμε για τη Γεωργία, η οποία έχει αναδειχθεί στον προτέτιο των προβλημάτων επειδή προκαλεί πολλές εκπομπές ή παράγει υπερβολικά ή υπερβολικά πολλά, υπερβολικά λίγα βιοκάψιμα κλπ. Εγώ έχω επιφυλάξει απέναντι στις παραγράφους 6 και 35. Ευχαριστώ και τώρα ο κύριος Φερέιρα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η συζήτηση όσον αφορά την προώθηση του εμπορίου και μάλλον την πρόθεση της ανάπτυξης μέσω του εμπορίου δεν μπορεί να παραβλέπει τις αρνητικές επιπτώσεις της ε, παγκοσμιοποίησης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ε, αντίθετα από τους, τους γενικούς κανόνες του ελεύθερου εμπορίου για αυτές τις χώρες ε, οι επιπτώσεις είναι περισσότερη φτώχεια, περισσότερη ενισότητα, περισσότερες δυσκολίες που επιβάλλονται στην διαφοροποίηση τη οικονομία του πλήρη ανεξάρτηση και μεγαλύτερη ε, απαλωτρίωση των ε, φυσικών πόρων. Ε, η ανάπτυξη μέσω του εμπορίου σημαίνει συμπληρωματικότητα, πολιτικές συνεργασίες για την ανάπτυξη, ιδιαίτερη προσοχή για την ανάπτυξη του Νότου και μια μεγάλη προσοχή στους όσους συνυπογράφουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση τις συμφωνίες οικονομικής συνεργασίας ώστε να είναι δίκαιοι στις χώρες τους γιατί οι συμφωνίες αυτές διαφορετικά είναι απλώς προς όφελος των πλούσιων και δεν βοηθούν τους πιο αδύναμους. Ευχαριστώ. Η κυρία Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στα πλαίσια του Διεθνούς Εμπορίου με τις Αναπτυσσόμενες Χώρες Θέλω να ρωτήσω ποια είναι η επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ποια είναι η θέση του εισηγητή σε σχέση με την αρχή της κυριαρχίας των τροφίμων που είναι ε, ένα καινούργιο συλλογικό ανθρώπινο δικαίωμα. Υπάρχει σχέση με τον ειδικό εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα τρόφιμα και την κυριαρχία των τροφίμων. Η ιδέα είναι προφανώς ότι κάθε χώρα ή κάθε κοινότητα ε, έχει το δικαίωμα να παράγει τα δικά της τρόφιμα και οι επιτόπιοι καταναλωτές έχουν το αντίστοιχο δικαίωμα πρόσβαση σε τοπικά παραχθέντα φρέσκα και υγιεινά τρόφιμα. Εμεί το τηρούμε αυτό το δικαίωμα της κυριαρχίας των τροφίμων ή όχι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μικολάσικ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι το διεθνές εμπόριο είναι από τους αποτελεσματικότερους τρόπους καταπολέμησης της φτώχειας και βελτίωσης της ε, οικονομίας των φτωχών χωρών και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, φροντίσει τους φτωχούς ε, στον κόσμο, αυτό σημαίνει ε, στρέβλωση των βασικών αρχών της. Ένας άμεσος τρόπος βοήθειας των λιγότερων προνομιούχων είναι το εμπόριο. Το εμπόριο ε, όμως, ε, ε, ε, υπ' αυτή την έννοια έχει κάποια προβλήματα. Δύο αναφέρονται στην έκθεση. Το ένα πρόβλημα είναι η διαφθορά και δεύτερον η στάση των πολιεθνικών εκτός συνόρων της Ένωση. Η Ένωση δεν μπορεί να στηρίζει διεφθαρμένα καθεστώτα και η επιλογή επιχειρηματικών εταίρων είναι ένας καλός τρόπος για την καταπολέμηση της διαφθοράς αλλού. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η εταιρική ευθύνη από τις πολυεθνικές που συμπεριφέρονται διαφορετικά στην Ευρώπη και διαφορετικά εκτός Ευρώπης. Ευχαριστώ. Τελευταίος ο μιλητής, ο κύριος ε, Κέλλη. Ε, αναμφίβολα το εμπόριο είναι σημαντικό για την ε, ευημερία της ανθρωπότητας και όλο και περισσότερο ακούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το εμπόριο ιδιαίτερα εις ό,τι αφορά την ανάπτυξη ε, συμφωνιών ελευθερών συναλλαγών. Οι περισσότερες αυτές οι εμπορικές συμφωνίες βελτιώνονται σύν χρόνο, καθώς η Κομισιόν αντιμετωπίζει τις δυσκολίε του παρελθόντος και επιτελεί προόδους και βελτιώσεις και γνωρίζει καλύτερα τι αντίκτυπο θα έχουν οι συμφωνίες στις χώρες με τις οποίες συναλλάσσεται ε, ε, πώς επηρεάζεται η πολιτική κατάσταση. Σίγουρα δεν μπορούμε να ανεχθούμε την διαφθορά, της πολυεθνικές κλπ. Όμως σε τελευταία ανάλυση γίνεται πρόοδος ε, σταδιακά και εκεί όπου υπάρχουν δυσκολίες στη Γεωργία οι ρήτρες αναθεώρησης είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης αυτών των καταστάσεων. Ευχαριστώ. Και τέλος για να ολοκληρώσει θα δώσω το λόγο στην Επίτροπο Κρούς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλω να ευχαριστήσω την ε, Επιτροπή και τον ε, εισηγητή, τον κύριο Σβένσον και την Επιτροπή Ανάπτυξη. Ο, ο, ο συνάδελφός μου, ο κύριος Στεκόχ, ε, λυπάται που δεν μπορεί να είναι εδώ για να συζητήσει για το θέμα αυτό της ανάπτυξης μέσω εμπορικών συναλλαγών ε, και οπωσδήποτε δεσμεύεται να, ε, δώσει, να ανταποκριθεί με βάση τις προτάσεις που έχουν γίνει στα πλαίσια της εντολής του. Ε, ιδιαίτερα θέλουμε να ε, δημιουργηθεί πολύπλευρο εμπόριο και πρόταση για μια συνεκτική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υπεύθυνη, τον υπεύθυνο χειρισμό των πόρων. Ε, που είναι σημαντικό. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια θέματα που αναφέρονται στην έκθεση ε, με τα οποία συμφωνούμε. Πρώτον, θετική συμβολή του εμπορίου και των επενδύσεων για την μεγέθυνση και την ανάπτυξη. Όπως λέει και η ανακοίνωση, καμιά χώρα δεν έχει επιτύχει μακροπρόθεσμη ανάπτυξη χωρίς άνοιγμα στο εμπόριο και αντίστοιχες συνοδευτικές πολιτικές και συστήματα διακυβέρνησης. Αυτό είναι ένα ξεκάθαρο ε, παράδειγμα ε, συνοχής της πολιτικής που θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερον, η εμπορική πολιτική επηρεάζει πολλούς εμπλεκόμενους. Αυτό που κάνει με τις εμπορικές συμφωνίες η Ένωση είναι να δημιουργήσει ένα προβλέψιμο μακροπρόθεσμο νομικό πλαίσιο που θα επιτρέπει όλων των ειδών της επιχειρήσης να συνεργαστούν με τρόπο βιώσιμο. Αυτές οι συμφωνίες είναι ισχυρά εργαλεία και ε, δημιουργούν πολλές προσδοκίες. Αυτό βέβαια από μόνο του είναι πολύ θετικό. Βέβαια, μια εμπορική συμφωνία από μόνη της δεν μπορεί να τα λύσει όλα τα προβλήματα. Ε, στις ε, διεθνείς ε, και εξωτερικές σχέσεις. Υπάρχουν λοιπόν θεσμικά όργανα που παρακολουθούν την εφαρμογή και επαναπροσδιορίζουν το πλαίσιο, το θεσμικό όταν χρειάζεται και κάθε εμπλεκόμενος έχει το ρόλο του. Οι τελωνιακοί, οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις, οι καταναλωτές και οι ενδιαφερόμενοι πολίτες. Η ε, κυρία Μόρβεϊ μίλησε για το θέμα της αλληλεγγύης στον τομέα των τροφίμων. Θα συζητηθεί αυτό στα πλαίσια του ΠΟΕ και συγκεκριμένα της Υπουργική Συνόδου στον Παλί τέλος του χρόνου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετέχει στις συνομιλίες αυτές. Θεωρούμε όμως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είχε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από αυτά που αναφέρονται στην έκθεση. Ε, η εμπορική πολιτική της Ένωσης ε, έχει σαφουφείς αναπτυξιακούς στόχους. Ε, είναι πολύ συγκεκριμένη η εμπορική μας προσφορά και λαμβάνει υπόψη της τα επιμέρους προβλήματα των χωρών στις οποίες απευθυνόμαστε. Επίσης είναι φιλόδοξη η πολιτική μας και διαπεριφερειακή. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα πρόγραμμα για να λάβουμε υπόψη μας την αλλαγή του κόσμου μετά τη δεκαετία του 70 όταν δώσαμε μερίς προτιμησιακές ε, ε, ε, εμπορικές και θεσμολογικές προτιμήσεις. Δεύτερον, επίσης αυτό ισχύει και για τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης που είναι ευέλικτες και ε, αντιμετωπίζει τις χώρες και ως οικονομίες ε, που ε, έχουν δυνατότητα έτσι να επιτύχουν. Εμείς κάναμε πολλές πρόοδους στις περιφερειακές διαπραγματεύσεις στα πλαίσια της εντολής μας και εξακολουθούμε να φιλοδοξούμε ότι θα ολοκληρώσουμε ε, πριν τελειώσει η θητεία της Επιτροπής σε πολλές ακόμα ε, συμφωνίες. Ως ε, Επιτροπή υπεύθυνη για την ψηφιακή οικονομία σας διαβεβαιώνω ότι η Αφρικανική Ήπειρος έχει αξιοποιήσει την τεχνολογία των κινητών τεχνολογιών με τρόπο που αποφέρει απτά και καινοτόμα ωφέλη σε όλους τους ανθρώπους. Εμείς την, την Αφρική έχουμε υπόψη μας ε, στις συμφωνίες μας. Και τέλος για τα ανθρώπινα δικαιώματα θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η πολιτική της Ένωσης διεξάγεται με πλήρη σεβασμό των αρχών και στόχων της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε και τώρα θα ήθελα να σας αναγγείλω ότι έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα εξαχθεί αύριο στις 12.